διαδικτύου. Εκ μέρους της Επιτροπής, ε, πρώτος ομιλητής, τον βλέπω, είναι ο Αντιπρόεδρος Άντρους Άντζιπ. Ε, μόλις καθίσετε έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ. Ε, η Επιτροπή καλωσορίζει την πρωτοβουλία το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο για την έγκριση ψηφίσματος για την ανανέωση ε, του Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Αυτό τονίζει πολύ σημαντικές πτυχές ε, της ε, παγκόσμιας συζήτησης για την διακυβέρνηση του διαδικτύου. Εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα αυτό το ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία για την βελτίωση του πολυσυμμετοχικού μοντέλου για την διακυβέρνηση του διαδικτύου θέμα πάρα πολύ σημαντικό για την κοινωνία αλλά και για την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, πέρυσι γκρίναμε την ανακοίνωση για την διακυβέρνηση του διαδικτύου και για την ε, σχετική πολιτική τον Νοέμβρη ακολούθησαν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για να τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του Παγκοσμίου Διαλόγου για το ζήτημα αυτό. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζονται στενά για τα θέματα αυτά, κυρίως στο, προ... στο πλαίσιο του φόρουμ ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου IGF, ε, κυρίως για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να συνεχίσει τις προσπάθειες σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο. Το σημερινό ψήφισμα είναι ένα ε, ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι και επίκαιρο το ζήτημα διότι το 2015 θα είναι ε, κρίσιμη σημασία σε έτος για την οικονομική διακυβέρνηση και έπονται πολύ σημαντικές ε, αλλαγές. Με τις νέες τεχνολογίες διαπιστώνουμε πόσο μεγάλη σημασία και μεγάλο αντίκτυπο έχουν οι συζητήσεις που γίνονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κοινός μας στόχος είναι να εξασφαλίσουμε πώς θα παραμείνει οικουμενικός πόρος ε, το διαδίκτυο και δεν θα χρησιμοποιηθεί από λίγους ε, που εξυπηρετούν συγκεκριμένα πολιτικά και οικονομικά ε, συμφέροντα. Το διαδίκτυο είναι κοινό αγαθό. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα που βασίζεται στη συνεργασία, στην εμπιστοσύνη και ξεκάθαρους κανόνες με τους οποίους θα υπάρχει συμμόρφωση. Έτσι θα νομιμοποιηθούν έτσι περαιτέρω οι κείμενες ρυθμίσεις για την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου. Πέρσι λήφθη απόφαση από ε, τις αρχές των ΗΠΑ για την μεταρρύθμιση, ε, για την ε, μεταβίβαση συγγνώμη, βασικών λειτουργιών για τα domain names των ΑΙΑΝΑ. Είναι γνωστό αυτό η μετάβαση ΑΙΑΝΑ και γιατί έδωσε τη συγκατάθεσή της για τη χρήση του πολυσυμμετοχικού μοντέλου. Ελπίζουμε ότι για τα λεπτότερα ζητήματα, όπως παραδείγμα χάρη αυτά που σχετίζονται με την λογοδοσία της ICAN θα δοθούν ικανοποιητικές απαντήσεις. Δεν μπορεί να λειτουργεί ως δικαστική αρχή το IGF όταν υπάρχουν νομικές διαφορές με άλλους εμπλεκόμενους φορείς. Ε, η βασική πρόκληση για το μέλλον είναι να υπάρχει αντιστάθμιση των εξουσιών και έλεγχος της λειτουργίας του δωρηνού συστήματος ε, από ε, πολλές πλευρές. Προς το παρόν θα εξετάσουμε τα πορίσματα της ε, παγκόσμιας διάσκεψης για την κοινωνία των πληροφοριών Ξέρουμε επίσης ε, ότι τα συμπεράσματα αυτά θα συζητηθούν και στο IGF. Υπάρχουν κάποια ανησυχητικά σημάδια, ανησυχητικές εξελίξεις ε, που παρεμποδίζουν ε, την πολύπλευρη αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων θα πρέπει να μερμήσουμε το σώστη η παγκόσμια διάσκεψη WSIS δεν θα οδηγήσει ε, σε ε, κυβερνητικό έλεγχο από πλευράς κάποιων κρατών μελών ε, του διαδικτύου. Χρειαζόμαστε ένα κρατεότερο IGF ως προς τη χρηματοδότηση αλλά και ως προς θέματα περιεχομένου. Είναι καταλητική σημασία σε αυτό ώστε να έχουμε την απαιτούμενη σταθερότητα για να καλύψουμε τις αυξανόμενες προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας. Επίσης ε, χρειαζόμαστε και άλλες πλατφόρμες ε, για να ολοκληρωθούν οι τωρινές συζητήσεις ε, για τα διάφορα ζητήματα διακυβέρνηση του διαδικτύου, χωρίς όμως να υπονομευθούν οι προσπάθειες που ήδη γίνονται ε, σε σχέση με τα αποτελέσματα του Net Mandial θα ήθελα να ανακοινώσω με μεγάλη χαρά ότι συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρωτοβουλία Net Mandial. Ε, θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την περαιτέρω ε, πύρωση του πολυσυμμετοχικού μοντέλου για, την οικονομική, για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Ας ακούσουμε τώρα τους εκπροσώπους, λέει ο των πολιτικών ομάδων, ε, Ντελικαστήγιο Βέρα. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Άνσιπ. Συζητούμε ένα ψήφισμα που στηρίζεται από την ε, στρεπτική πλειοψηφία του Ευρωκοινοβουλίου και υπάρχει ένας πολύ σαφής στόχος εδώ. Ε, ο βασικός στόχος, πέραν όλων των υπολείπων βεβαίω, είναι να περάσει επιτέλους ένα μήνυμα. Το ε, φόρουμ για την διακυβέρνηση του διαδικτύου να συνεχίσει να εργάζεται και να εξακολουθήσει τη δράση του. Κάτι πολύ σημαντικό για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια του 2015. Ε, θα ανανεωθεί τότε η εντολή ή όχι. Αυτό είναι το ερώτημα και θα πρέπει το Ευρωκοινοβούλιο να προωθήσει τη δράση του φόρουμ αυτού βάσει των εμπειριών που είχαμε και συνεργαζόμενοι ως τώρα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει να φροντίσουμε ακριβώς αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί για να παραταθεί και η εντολή και στη διακυβέρνηση του διαδικτύου να υπάρξει απαραίτητη ασφάλεια. Διότι ε, η απειλή για αυτή την ασφάλεια είναι ότι οι διακυβερνητικές δράσεις δεν αρκούν. Χρειάζεται ε, να ε, υπάρξει μια πολυμερής προσέγγιση που να οδηγήσει σε μια σφαιρική αντιμετώπιση. Γι' αυτό ζητούμε ένα σαφές μήνυμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο εκ μέρους των κρατών μελών να υποστηρίξουν την ε, την ε, δράση αυτή για να ανανεωθεί η εντολή του διακυβερνητικού φόρου. Εκ μέρου των Σοσιαλδημοκρατών, για δύο λεπτά η κυρία Καμέρα Φεύερτα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, οι εκπρόσωποι 120 ε, χωρών ε, πήγαν στην Κωνσταντινούπολη και δήλωσαν τι είναι ακριβώς αυτό το φόρουμ ότι υπάρχει δυνατότητα χρήσης του ίντερνετ και να έμπνευση της συζήτησης για το θέμα αυτό. Η εντολή του ε, Κοινοβουλίου είναι να έχει εφαρμογή του, άρθρου, ε, του σχετικού άρθρου για τα ανθρωπίνα δικαιώματα που ασχολείται με το διαδίκτυο. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να το ε, τηρούμε. Η διακυβέρνηση στο διαδίκτυο είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Θα πρέπει να βρούμε τα προβλήματα, τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ως τώρα το Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός είχε θέσει αυτό το θέμα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είχαμε εκπρόσωπους από χώρες οι οποίοι ε, θεωρούν ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε συγκέντρωση της ε, ισχύω ε, και να υπάρχει παραβίαση δικαιωμάτων τελικά. Πρέπει λοιπόν ε, να ε, διασφαλίσουμε την ουδετερότητα. Η ΕΠΑ πολύ συχνά αναγνώρισε τα σημάδια των καιρών και ο επικεφαλής του FCC μίλησε για την ξεκάθαρη ουδετερότητα την οποία θα, έχουμε και στην, θα πρέπει να έχουμε και στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σταματήσει το μπλοκάρισμα ή η αργή επεξεργασία δεδομένων. Ε, δεν θα πρέπει να πέσουμε λοιπόν στη ρητορική ε, αυτών που λένε ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός. Ναι, λειτουργεί, αλλά θα πρέπει ε, να έχουμε τις δυνάμεις ελεύθερες γιατί είναι πολύ σημαντικό ε, όλες οι δομές ε, να βοηθήσουν στην ελευθερία της επικοινωνίας. Ε, γι' αυτό θεωρώ ότι η πλατφόρμα του φόρουμ αυτού είναι πολύ σημαντική για την ελευθερία στο ίντερνετ. Ευχαριστούμε πολύ εκ μέρου ε, των ε, Ευρωπαίων Συντηρητικών η Βίκη Φόρτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Το διαδίκτυο πρέπει να είναι ελεύθερο αλλά και ασφαλέ. Να υπάρχει πρόσβαση για όλου αλλά και χωρί προπολικό κόστο. Να είναι συναρπαστικό, δυναμικό και ποικιλόμορφο. Στην Ευρώπη έχουμε ξεκινήσει από μια πολύ καλή θέση. Και με το Παγκόσμιο Φόρουμ έχουμε δει ποιε είναι οι χώρε που τεχνολογικά είναι προηγμένε. Οι πρώτε τρει είναι στην Ευρώπη. Όμω το ε, δυναμικό που δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πρέπει να αξιοποιηθεί αν εφόσον κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα πρέπει οι πολίτε να ξέρουν ότι τα δικαιώματά του γίνονται σεβαστά και ότι τα δεδομένα ε, τα επεξεργαζόμαστε με υπευθυνότητα. Θα πρέπει οι επενδυτέ να γνωρίζουν ότι εμεί οι, οι πολιτικοί δεν θα αλλάζουμε διαρκώ του κανόνε που επηρεάζουν τι επενδύσει του και οι επιχειρήσει πρέπει να γνωρίζουν να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ίσοι κανόνε παιχνιδιού όταν οι μικρότερε επιχειρήσει δεν ε, μπλοκάρονται από τι μεγαλύτερε ούτε οι νεότεροι επενδυτέ από του παλιού. Η απελευθέρωση του διαδικτύου είναι απαραίτητη. Πρέπει να έχουμε τεχνολογική ευδετερότητα, να την εξασφαλίσουμε και να φροντίσουμε να μην πρόκειται φραγμοί για μελλοντικέ επενδύσει Και για την, ε, για την προστασία του ιδιωτικού βίου. Δεν θα πρέπει να υπονομεύσουμε την ασφάλεια των κοινωνιών μα και των παιδιών μα, Τηρώντας δεδομένα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι δεν θα επιβάλλουμε υπερβολικό άχθο στι μικρέ επιχειρήσει η κοινωνία να αξιοποιήσει την δημιουργία μεγάλων τραπεζών δεδομένων θα πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι προστατεύονται τα θεμέλια δικαιώματα, ναι μεν, αλλά από την άλλη και η, ασφάλεια, η βασική ασφάλεια απειλείται και γνωρίζει πιέσει. Θα πρέπει λοιπόν να δεχτούμε συμβουλέ από εμπειρογνώμονε, να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μα, αλλά να προβλέψουμε και τα μέσα για να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πολιτών. Για να ε, λάβει σάρκα και ωστά αυτό το όραμα, θα πρέπει να ε, καταβάλουμε μεγάλε προσπάθειε όλη την Ευρώπη, συνεργαζόμενοι με του βασικού μα εταίρου, προστατεύοντα του καταναλωτέ και τι επιχειρήσει, το κοινό και τι δημόσιε αρχέ. Και ελπίζω ότι θα μα βοηθήσει το Παγκόσμιο Φόρουμ να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία και ότι όλα θα πάνε καλύτερα εφόσον συνεργαστούμε εντατικά. Ευχαριστούμε κυρία Φόρντ. Επόμενος, η κυρία Κάλλας για τους ε, ε, ε φιλελεύθερους. Ευχαριστώ Στη συζήτηση αυτή διερωτόμαστε αν το διαδίκτυο είναι μεταξύ των θεμελιωδών δικαιωμάτων, αν είναι ένα αγαθό κοινό όπως το νερό. Εάν έτσι είναι, ποιοι είναι οι κανόνες ε, για το διαδίκτυο. Πρέπει σε όλη αυτή τη συζήτηση να θυμόμαστε ότι το διαδίκτυο δεν είναι εθνικό ή ευρωπαϊκό. Σε αυτό το παγκόσμιο, στην παγκοσμιοποιημένη αγορά, οι κανόνες ε, της ε, εμπορίας και της πρόσβασης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και στην πρόσβαση στο διαδίκτυο. Γι' αυτό εμείς Ευρωπαίοι πρέπει να στηρίξουμε και να συμμετάσχουμε ενεργά στο Παγκόσμιο Φόρουμ του γιατί υπάρχει αυτή η συζήτηση σε διεθνέ επίπεδο για το διαδίκτυο, τι προκλήσει που θα μα αναγκάσει να αντιμετωπίσουμε και τι βασικέ ανάγκε που δημιουργεί. Εκ μέρου των φιλελευθέρων έχω τονίσει στο ψήφισμα αυτό ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδει ελευθερίε που έχουμε ε, εκτό διαδικτύου θα πρέπει να γίνονται σεβαστέ και ε, στο διαδίκτυο. Αυτό ε, πρέπει να ε, ισχύσει μαζί με την αποφυγή της μαζικής παρακολούθησης πολιτών αλλά και της κρατικής παρακολούθησης του διαδικτύου. Αυτά αντίκεινται με τις βασικές μας ελευθερίες στη χώρα μου, την Εστονία. Ε, καταλάβαμε τη δεύτερη θέση για την ελευθερία στο διαδίκτυο στην παγκόσμια κατάταξη, αλλά ήμασταν μάλλον εξαίρεση, καθώς 84% των χωρών είχαν το 2014 πολύ αδύναμους νόμους ή καθόλου νομοθεσία για την προστασία των πολιτών κατά της μαζικής παρακολούθησης. Και τα πράγματα χειροτερεύουν. Χειροτερεύουν γιατί το 64% ε, ήταν το ποσοστό του 2013. Ε, να σταθούμε σε ένα σημείο λοιπόν. Τα δικαιώματα των ε, πολιτών για ασφαλείς επικοινωνίες, ακόμη και με την κρυπτογράφηση των στοιχείων τους, είναι στοιχεία που θα πρέπει να τα δει και το Παγκόσμιο Φόρουμ. Νομίζω ότι ο ιδιωτικός βίος των πολιτών δεν θα πρέπει να απελευθερωθεί. Δεν μπορεί το διαδίκτυο να είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα έκφρασης και ανταλλαγή ιδεών χωρί την προστασία του ιδιωτικού βίου. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υπάρξει ενεργή στην προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών και σε διεθνέ επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενο ομιλητή, ο κύριο Ρέιμον, εκ μέρου ε, των Πρασίνων. Δυόμιση λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ίντερνετ με μια σημαντική αντίφαση. Είναι πάρα πολύ ρυθμισμένο το ε, σύστημα του ηλεκτρονικού ε, υπολογιστή, όμως θέλουμε ε, να, θέλω να πω ότι πρόκειται για τεχνικούς κανόνες. Στην ουσία δεν μπορεί να ελέγξει την, η ιστορία των πολιτών που θα πρέπει να έχει ελεύθερη, τη δυνατότητα ελευθερίας παγκόσμια ιστορία έτσι έγινε όπως είναι σήμερα. Αυτή η ελευθερία λοιπόν που έχει τεχνητά ρυθμιστεί τώρα λοιπόν να απειλείται λόγω των συμφερόντων διότι οι κυβερνήσεις ε, και οι εταιρείες προσπαθούν ε, να ενισχύσουν αυτή τη ρύθμιση του ε, διαδικτύου και να έχουν από αυτό όφελος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να συμμετέχει σε αυτό το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου έτσι ώστε να βοηθήσει σε διεθνέ επίπεδο να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια κατά τη υπερβολική ρυθμίση. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, είναι πολύ σημαντικό που αυτό το ψήφισμα έχει ε, μεγάλη πλειοψηφία γιατί υποστηρίζει την οδετερότητα στο θέμα ας πούμε, της παρακολούθησης. Το ε, δίκτυο χρειάζεται οδετερότητα και ελπίζω όταν θα ψηφίσουμε να έχουμε καταφέρει να φτάσουμε τουλάχιστον στο μισά του δρόμου για τον ορισμό της ουδετερότητας γιατί πραγματικά δεν κατανοούμε θεωρώ ε, τι ακριβώς είναι αυτή η ουδετερότητα ότι υπάρχουν επίπεδα ε, δεν μπορούμε όμως να την κατακαιρματίσουμε ε, θα πρέπει όλοι να έχουν ισότιμη μεταχείριση και ε, να μην υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Έτσι λοιπόν ε, θα έλεγα ότι πρέπει να μιλάμε για προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των πολιτικών δικαιωμάτων και προστασία κατά της παρακολούθησης έτσι ώστε στο μέλλον το δικαίωμα της ελευθερίας ε, του λαού ε, να ε, μην υπονομεύεται αμέσα από παρακολουθήσεις και για τα συμφέροντα των μυστικών υπηρεσιών. Τέλος, να ζητήσω το εξής. Όταν εμείς ως κοινοβούλιο θέλουμε να συμμετέχουμε σε αυτό το φόρουμ, καλό θα είναι να έχουμε όσο μεγαλύτερη εκπροσώπηση γίνεται με όσο περισσότερα μέλη στην Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, εκ μέρους του EFTD για δύο λεπτά. Αν ε, ε, υπάρχει μια φράση που θα πρέπει να μας κάνει να ε, είμαστε ναι, με επισταμένη την προσοχή μας είναι ότι ε, το ίντερνετ ε, πρέπει να έχει διακυβέρνηση. Ε, το θέμα του IGF τα τελευταία χρόνια ήταν γεμάτο με λέξεις κλειδιά και ηχηρές λέξεις. Όμως η ίδια η ύπαρξη του ίντερνετ, η οποία είναι ανταλλαγή ιδεών ελεύθερη στην ουσία τρομοκρατεί τα κράτη που δεν μπορούν πλέον να το ελέγξουν γιατί το ίντερνετ είναι κατά της καθεστικίας ε, τάξης ε, γιατί ε, υπάρχουν ας πούμε προσπάθειες όπως η έκδοση της βίβλου την καθομιλουμένη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα θέσουμε στο προσκήνιο ε, και θα πρέπει να ε, σταματήσουμε ε, την παιδική πορνογραφία ή τις πράξεις του τρομοκρατίας. Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε ότι το ίντερνετ έχει να κάνει με τη δημιουργία ελεύθερων επιχειρήσεων. Αν η κυβέρνηση, όταν ακούμε ότι η κυβέρνηση θέλει να προωθήσει την ελεύθερη επιχειρηματικότητα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να το κάνουν αυτό και αν λέμε ότι αυτές θα οδηγήσουν στην καινοτομία θα πρέπει να ξέρουμε ότι αυτό είναι ε, μία παρέστηση. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ε, όρους ε, που θα μας βοηθούν στο να έχουμε καινοτομία και όχι να θολώνουμε τα νερά. Θα πρέπει να έχουμε διεθνή στάνταρ, τα οποία όμως πρέπει να τα κάνουμε με βάση πολλή εργασία, αλλά θα πρέπει να αφήσουμε και τους ανθρώπους να δράσουν ελεύθερα. Ευχαριστώ κύριε Γιάλ, ο κύριος Γιάλ για ένα λεπτό. Σήμερα έχουμε ένα θαυμάσιο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη, την πολιτιστική, την ιδεολογική και την πολιτική μα έκφραση. Εδώ πρέπει να αναζητήσουμε ζώνε ελευθερία για το μόνο πραγματικό δημοκρατικό κεκτημένο των τελευταίων 15 ετών. Είναι το τελευταίο μα επίτευγμα. Πρέπει λοιπόν η τεχνική ιεραρχία και η ιεράρχηση που χαρακτηρίζει την Επιτροπή μας να μην εμποδίσει την έκφραση στο διαδίκτυο των διαφόρων δευμάτων της ε, ζώσας κοινωνίας. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο αυτή η άειλη τεχνολογία που ε, δεν ε, ε, επιτρέπει στην παγκοσμιοποίηση να παραμείνουν ακλόνητες οι προκαταλήψεις του παρελθόντος να έχει την ε, σωστή διέξοδο. Θα πρέπει λοιπόν η ε, κατάργηση στο τόπο όπως η τζιχαντιστική να, οι ισλαμιστικές ακραίες εκφράσεις όλα αυτά να τα δούμε στο πλαίσιο της σωστής διάρθρωσης διότι θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τις μόνιμες εξαιρέσεις που μπορεί να ήταν επιζήμιες για όλους. Θα πρέπει η δημοκρατία δημοκρατικές ελευθερίες των πολλών να μην ε, ε, ε, καταργώνται, γιατί για να αποφύγουμε τα αεροπορικά δυστυχήματα δεν πρόκειται να καταργήσουμε την αεροπλοεία, δεν ήταν λογικό κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ κυρία Φερχαέν για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το 2015 θα είναι πολύ σημαντικό για την δημιουργία νέων δομών στη διακυβέρνηση του ίντερνετ. Σε αυτή τη διεθνή συζήτηση η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμετέχει εντατικά. Το IGF στο παρελθόν είχε μια επικοδομητική συμβολή με ένα πλαίσιο για διεθνεί ανταλλαγέ όπου συμμετείχαν όλοι όσοι συμμετείχαν κάθε είδου συμφέρον. Στο μέλλον λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια επιμήκυνση αυτή τη εντολή. Και είναι σημαντικό ιδιαίτερα να τονίσουμε τη σημασία ε, της πολυσυμμετοχικής αυτής δράσης στο IGF. Είναι πολύ σημαντικό να ε, έχουμε ανταλλαγή απόψεων για να μπορέσουν να βρεθούν πάρα πολύ σημαντικές και εφαρμόσιμες λύσεις για αυτό το θέμα η διακυβερνητική ε, διάσταση δεν θα πρέπει να σταματήσει υπέρ των μικρών ομάδων. Θέλουμε ε, να έχουν ε, συμμετοχή όλοι όσοι εκπροσωπούν διάφορα συμφέροντα έτσι ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η η στάση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και να μπορούμε να έχουμε πραγματική ε, δουλειά η οποία θα μπει στην πράξη για αυτό το θέμα. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ξέρουμε ότι η οργάνωση του διαδικτύου είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να προωθήσουμε την ε, διεθνοποίηση χωρίς ε, να μην μένουμε πίσω για τα διάφορα συμφέροντα. Θα πρέπει να υπάρχει λογοδοσία και διαφάνεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να γνωρίζουμε και για τη λειτουργία η ΕΕ που και αυτή οδηγεί στη διεθνοποίηση και πρέπει να προωθηθεί. Θεωρώ και εδώ ότι πρέπει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο να δράσουν και συμφωνώ με αυτό που είπε ο συνάδελφος να στείλουμε μια πιο ισχυρή αντιπροσωπεία στην επόμενο φόρουμ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ευχαριστώ. Επόμενος ε, ε, ο μιλητής ο κύριος Πόχεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που έχει ηγετικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτό τον ε, κρίσιμη σημασία ε, τομέα. Το 2015 ε, έχει ιδιαίτερη σημασία όχι μόνο λόγω της παράτασης εντολής του IGF αλλά και λόγω της μεταβίβασης της εκχώρησης αρμοδιοτήτων για την παραχώρηση αριθμών και για τα domain names σε διεθνή φόρα. Ε, όπως και άλλα μέλη της διεθνούς κοινότητας ε, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να παραταθεί η εντολή του Διεθνούς Φόρουμ για την Διακυβέρνηση διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ο διάλογος ε, να γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο λόγω και τη σημασία που έχει για την οικονομία. Είναι πάρα πολύ σημαντικές συστάσει που απορρέουν από το IGF για θέματα ε, κανονιστικά, για θέματα προστασία τη ιδιωτική ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το φόρουμ και πρέπει να παραταθεί η εντολή του. Ευχαριστούμε. Η κυρία Καραντσόβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτω με τα σχόλια που έχουν γίνει μέχρι στιγμή, Ναι, πρέπει να ζητήσουμε παράταση εντολή του IGF και ναι θα πρέπει να συνεχίσουμε ε, σε αυτήν την άγουσα, δηλαδή ε, παγκόσμια να ε, μεταρρυθμίσουμε το τεχνικό πλαίσιο για την διακυβέρνηση του διαδικτύου. Η ψηφιακή αγορά είναι και θα παραμείνει το κέντρο της οικονομίας. Η ανάπτυξη από αυτό το τομέα ανέρχεται στο 11% και για το ΑΕΠ από το 3,8% θα περάσουμε στο 5,7% το 2016, ποσοστό δηλαδή του ΑΕΠ που αντιστοιχεί στο διαδίκτυο. Επίσης βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το τομέα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κανονιστική ρύθμιση στο διαδίκτυο σε θεσμούς που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ε, να μην ξεχνάμε ότι είναι δίκοπο μαχαίρι όμως οποιαδήποτε ε, εξέλιξη στο ρόλο που έχουμε, διότι υπάρχουν και κράτη που ε, δεν σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και πρέπει να επιδιώξουμε ε, η παγκόσμια διεθνή κοινότητα να παραμείνει ενωμένη κατά αυτών των κρατών μελών, κατά της λογοκρισίας, ε, κατά της παρεμπόδισης του δικαιώματος πληροφόρησης και της ελευθερίας έκφρασης ε, για να αποφύγουμε την μαζική παρακολούθηση και τα εμπόδια στο διαδίκτυο. Μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί η ανθρωπότητα να προχωρήσει. Σας ευχαριστούμε κυρία Καράντσοβα, η κυρία Ρέντα. Ένα λεπτό. Κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ίντερνετ είναι παγκόσμιο από τη φύση του. Παρόλο που το φόρουμ διακυβέρνηση του δικτύου δεν λαμβάνει αποφάσεις, έχει γίνει σημαντικό κομμάτι του παγκοσμίου διαλόγου για αυτό το θέμα. Πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να διασφαλίσουμε ότι όλοι θα συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο με λογικό τρόπο. Η κοινωνία των πολιτών, οι κυβερνήσει, οι εταιρείε, όλοι συμμετέχουν στο φόρουμ. Αυτέ οι ομάδε πολλέ φορέ πρέπει να ε, βασιστούν περισσότερο ε, στην εξωτερική υποστήριξη. Ας πούμε, η κοινωνία των πολιτών πρέπει να υποστηριχτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει σταθερή χρηματοδότηση για να υπάρχει ανεξαρτησία σε πολιτικό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να δούμε τι έγινε στην Κωνσταντινούπολη. Υπήρχαν τοπικές ομάδες της αντιπολίτευσης που είπαν ότι δεν είχαν ε, συμπεριληφθεί και έκαναν ένα άλλο παράλληλο φόρουμ για να ακουστούν. Ε, είναι λοιπόν ε, σημαντικό ε, να ακουστεί ότι υπάρχει αυτή η αντιπολίτευση των εισαγωγικών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δώσει χρηματοδότηση αλλά να επιτρέπει σε όλες τις πολιτικές ομάδες να στέλνουν εκπροσώπους στο φόρουμ για να υπάρχει πλήρης εκπροσώπηση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τροσίνσκι για ένα λεπτό. κυρία, κυρία Τροσίνσκι, ευχαριστώ Πρόεδρε, όντω στο διαδίκτυο υπάρχει πραγματική έκφραση ελευθερία που πρέπει να διατηρηθεί. Όμω με τα προγράμματα μαζική παρακολούθηση από τι μυστικέ υπηρεσίε των ΗΠΑ υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι για την εσωτερική ασφάλεια και την ανεξαρτησία των πολιτικών των κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πρωτίστω και οι ευρωπαϊκοί λαοί περιμένουν μια ισχυρή αντίδραση και χωρί ε, αμφισημία από την πλευρά σα. Θα πρέπει να ικανοποιήσετε το αίτημα αυτό με την ανανέωση τη εντολή του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Διαδίκτυο. Η διεθνή διακυβέρνηση του ε, διαδικτύου είναι ε, καθοριστική σημασία γιατί τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει με διαφανή τρόπο να προστατεύονται καθώ και οι πόροι του ίντερνετ να αξιοποιούνται και να διατίθενται σε όλου με τον ίδιο τρόπο. Ε, θα πρέπει η αμερικανική προοπτική τη διακυβέρνηση πρέπει να αμφισβητηθεί με την έννοια ότι εμεί θα πρέπει να καθορίσουμε τη δική μα προοπτική. Θέλετε να υπάρχει κατασκοπία και να μπορούν οι ΗΠΑ να κάνουν ό,τι θέλουν από τη δική του πλευρά. Μονομερό. Έχουμε πολλέ λοιπόν, πολλού ενδιασμού ότι έχετε σκοπό να ε, προστατεύσετε τα δικά μα συμφέροντα και όχι αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών. Και με το ψήφισμα των πολιτικών ομάδων δεν υπάρχει κανένας, ε, καμία ανακούφιση, καμία ε, κάτι που να μας πείθει ότι οι Αμερικανικές αρχές δεν θα συνεχίσουν τη δράση τους. Πρέπει και η ευρωπαϊκή απάντηση να υπάρξει στο Παγκόσμιο Φόρουμ. Ευχαριστούμε η κυρία Τούνεν Χόενστάιν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε το Παγκόσμιο Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου είναι η πλέον δημοκρατική δομή που ε, διεξάγει συζήτηση για την, ε, διεξάγει μάλλον συζήτηση για, την, για, το, για το μέλλον του διαδικτύου συνολικά. Οι εταιρείε, οι εμπορευόμενοι, οι ομάδε πίεση, οι πολίτε, όλοι εκπροσωπούνται και η συζήτηση αυτή για το μέλλον του διαδικτύου είναι καθοριστική σημασία στη σήμερα ημέρα. Διότι έχει να κάνει με όλε τι προκλήσει που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Το διαδίκτυο είναι μια δυναμική ε, δομή. Οι χρήστε του περνούν όλο και περισσότερο χρόνο ε, με τις διάφορες εφαρμογές που διατίθενται, με την ε, χρήση των ε, εργαλείων έρευνας, αναζήτησης μάλλον. Εδώ πέρα υπάρχουν όλο και, υπάρχουν όλο και περισσότερες εφαρμογές που διατίθενται στους πολίτες για να καλύψουν τις ανάγκες τους και βεβαίως ανάλογα με τις ε, συσκευές, τις κατηγορίες συσκευών που πολλές φορές δεν είναι συμβατές μεταξύ τους. Αυτό, ε, αυτή η προσέγγιση σε κουτάκια κάνει το διαδίκτυο όλο και λιγότερο ελεύθερο και ανοιχτό. Αυτό είναι μεγάλος κίνδυνος από την άποψη και την προοπτική των χρηστών. Το διαδίκτυο πρέπει να απελευθερωθεί. Είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό η εντολή του Παγκόσμιου Φόρουμ για το Διαδίκτυο πρέπει να ανανεωθεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μια ιστορική επιταγή. Στην αρχή του 20ου αιώνα είχαμε την αρχή της αυτοκινητοβιομηχανίας. Ε, ε, τώρα ε, Έχουμε το φόρουμ, το οποίο είναι ένα ε, χώρος συζήτησης ε, για ένα ακόμα πιο ιστορικό θέμα. Είναι πολύ σημαντική η συμβολή του διαδικτύου και στην ιδιωτική ζωή και ε, θα πρέπει να έχουμε προστασία των προσωπικών δεδομένων και από την παρακολούθηση από τις μυστικές υπηρεσίες. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σωστή οργάνωση του διαδικτύου, το οποίο είναι ένα ανοιχτό ε, ε, κοινό αγαθό και θα πρέπει να παραμείνει έτσι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, εδώ στο Κοινοβούλιο να λαμβάνουμε αντίστοιχες αποφάσεις και ελπίζουμε ότι και το Συμβούλιο θα κάνει το ίδιο. Ευχαριστούμε πολύ. Επόμενος, ε, η επόμενη κυρία Σφαλκή. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διακυβέρνηση στο διαδίκτυο είναι αντίφαση από μόνη της, γιατί όλοι θέλουμε ένα παγκόσμιο ίντερνετ που θα είναι ανοιχτό, χωρίς ε, φραγμούς που δεν χρειάζονται. Όμως ε, θα πρέπει να ληφθούν πολλές αποφάσεις σε πολλά επίπεδα με το σωστό τρόπο για να γίνει αυτό και το πολυσυμμετοχικό μοντέλο θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο νόημα στην εποχή μας. Η ευρωπαϊκή ηγεσία δεν θα πρέπει να αφήσει τη διακυβέρνηση στη Ρωσία και στην Κίνα και σε άλλες χώρε που οι κυβερνήσει του ε, παίρνουν νομιμοποίηση και ε, ε, το φόρουμ θα πρέπει στην ουσία να απομονώσει τέτοιες ε, δράσεις. Θα πρέπει εμείς εδώ να διασφαλίσουμε την ουδετερότητα ε, στο χώρο μας αλλά και παγκοσμίω. και θα πρέπει να το κάνουμε αυτό προς όφελος των χρηστών, των μη κυβερνητικών οργανώσεων και όλων όσοι μπορούν να βοηθήσουν ώστε τα δικαιώματα να εφαρμόζονται και online και offline. Θα πρέπει λοιπόν το ίντερνετ να έχει ωφέλη για όλους μας και τώρα και στο μέλλον. Και αυτό να το διασφαλίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Σάκε. Έχουμε καλά για κάρτα από την κυρία Μορβάη. Δέχεστε. Κυρία Μορβάη, 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Συνάδελφε, είπατε και αναφέρατε την ε, βαλκανοποίηση και την καταστολή της ε, Ρωσίας ε, ως προς το διαδίκτυο. Για τον Έντουαρτ Σνόντεν που αποκάλυψε την παρακολούθηση από τις Αμερικανικές Αρχές στο διαδίκτυο και τώρα διαμένει στη Ρωσία. Τι έχετε να πείτε. Εκεί κατέφυγε για να συνεχίσει τη δουλειά του. Πώς το εξηγείτε. Πώς τα συνδυάζετε αυτά τα δύο. Uh, όπως τα γνωρίζετε συνάδελφε, επειδή ακριβώς ένας από αυτούς που αποκαλύπτουν πληροφορίες ε, ανέφερε τις καταχρήσεις των Αμερικανικών αρχών και των μυστικών υπηρεσιών του. αυτό δεν δικαιολογεί την καταστολή των δημοσιογράφων και την ελευθερία της εκφρασής τους από το Κρεμλίνο όταν θέλουν να εκφραστούν στο διαδίκτυο ή εκτός. Επιπλέον η Ρωσία ε, ζητά την ε, τήρηση δεδομένων και την αποθήκευσή τους στη Ρωσία. Αυτό βλάπτει την ελευθερία στο διαδίκτυο, όπως γνωρίζουμε όχι μόνο για τους Ρώσους πολίτες αλλά για τους ε, χρήστες του διαδικτύου διεθνώς. Ευχαριστούμε. Ε, θα πρέπει να διαφυλάτονται τα δικαιώματα έκφρασης, ελευθερίας έκφρασης στο διαδίκτυο, όμως υπάρχει και το δικαίωμα λήθης, ε, βασικό δικαίωμα για την προστασία των ατομικών δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα κατοχυρώθηκε το 2014, 13 Μαΐου, με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Οποιοςδήποτε βλάπτεται από πληροφορία που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο μπορεί να αποταθεί ε, στον διακομιστή για διαγραφή των στοιχείων ε, μετά την πάροδο ε, μιας εύλογης προθεσμίας ε, πολλών ετών. Καλό αυτό, αλλά δεν επαρκεί. Προσπαθεί να αντισταθεί η Google. Στις 6 Φεβρουαρίου του 2015 δημοσίευσε μία έκθεση ε, που αμφισβητεί αυτό το δικαίωμα αληθισία και γι' αυτό το φόρουμ για την διαδικτυακή διακυβέρνηση θα πρέπει επιγόντως να ασχοληθεί με τρία ζητήματα. Πρώτον, η προθεσμία ε, μετά την εκνοή της οποίας ε, μπορεί να υπαχθεί κάτι αυτό το δικαίωμα αλήθης. Δεύτερον, το πώς σχετίζεται αυτό με το δικαίωμα ενημέρωσης του κοινού και τρίτον, αν θα πρέπει πρέπει να υπάρχει έξτρα ευρωπαϊκή διάσταση αυτού του δικαιώματος για να αντιταχθούμε στο μοντέλο Google ε, των Αμερικανών. Σας ευχαριστούμε. Κυρία Νίπλερ, 1,5 λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Επίτροπε, συνάδελφοι. Χρειαζόμαστε ένα ε, διαδίκτυο στο οποίο θα έχουν όλοι πρόσβαση, δεν θα υπάρχουν διακρίσεις, ε, να πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στο διαδίκτυο, ότι υπάρχει προστασία των δεδομένων και της πνευματικής ιδιοκτησίας. Εδώ οι Ευρωπαίοι ε, ηθήνοντες ε, ε, θα πρέπει να λαμβάνουν μέρος σε αυτό το φόρουμ διότι είναι μια πολύ σημαντική πλατφόρμα και στο παρελθόν ε, μπόρεσε να εκπληρώσει τα καθήκοντά του. Θεωρώ λοιπόν και ελπίζω ότι η εντολή θα επιμηκυνθεί, θα παραταθεί και ε, όταν αυτό γίνει εμείς ως Ευρωπαίοι θα είμαστε μια ισχυρή φωνή διότι πρέπει να ακουστεί η φωνή μας και πρέπει να υποστηρίξω αυτό που είπε και η συνάδελφος Φερχάιν ότι πρέπει να έχουμε μια ισχυρή παρουσία μέσα από το Κοινοβούλιο ε, και μες και γι' αυτό ζητώ από τον Επίτροπο να φροντίσει γι' αυτό. Επίσης, να εδράτω με τις ευκαιρίες να σας θυμίσω ε, ότι υπάρχει η πρόθεση ενός ε, νομικού πλαισίου για τα καθήκοντα που έχουν να κάνουν με το διαδίκτυο και ζητώ από τον Επίτροπο να εξετάσει το θέμα της προστασίας των δεδομένων μέσα στα πλαίσια του πακέτου των τηλεπικοινωνιών έτσι ώστε να έχουμε πρόοδους και σε αυτό το θέμα, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις ε, διότι έτσι θα μπορέσει η Ευρώπη να κάνει τη δουλειά της και να έχει μια ισχυρή θέση σε διεθνές επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Δάντη, για ένα λεπτό. Αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το ίντερνετ είναι ένα, μια ανεξάτηλη δεξαμενή γνώσης. Μπορείς ε, να διαδώσεις ε, πληροφορίες, να δημιουργήσεις οικονομική ανάπτυξη και να έχεις και μια γεωπολιτικο-στρατηγική προσέγγιση. Ε, είναι μια νέα αγορά για μας η αυξανόμενη σημασία όμως του ίντερνετ πρέπει να συνοδεύεται και από επαρκείς εγγυήσει για τη διακυβέρνηση, για τη διαφάνεια, για την ασφάλεια και την ουδετερότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν ηγετικό ρόλο στον κόσμο έτσι ώστε να καλύψουμε το χαμένο χρόνο και να κάνουμε το διαδίκτυο πιο συμμετοχικό, πιο ασφαλές και ε, να του επιτρέψουμε να προστατεύσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες οι πολίτες πρέπει να εμπιστεύονται τα ψηφιακά περιβάλλοντα, θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν πλήρως τις νέες ευκαιρίες όπως το ηλεκτρονικό εμπόριο και τόσες πολλές ευκαιρίες που μπορεί να προσφέρει το δίκτυο. Το να έχουμε μια συμφωνία για την ασφάλεια ε, των ε, δικτύων πληροφορίες είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προ τα μπρο. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Σαλίνη για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σαλίνη, συγγνώμη. Ε, κύριε Επίτροπε, η ευκαιρία που έχουμε μέσα στα πλαίσια αυτού του φόρουμ διακυβέρνηση του διαδικτύου να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα φόρουμ όπου η κοινωνία μπορεί να κατανοήσει εκ νέου τον εαυτό της είναι ενώπιόν μας. Μέσα στο ε, ίντερνετ μπορούμε να έχουμε αρκετό χώρο για να αναπτυχθούν αξίες, ε, για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ε, στην προώθηση της εμπιστοσύνης ότι το δίκτυο θα μας επιτρέψει να, να προχωρήσουμε. Δεν είναι μόνο θέμα ασφάλειας, πρέπει να... Δεν συμφωνώ με όποιον λέει ότι σήμερα η έννοια της διακυβέρνησης είναι ασύμβατη με την έννοια του διαδικτύου και της ασφάλειας. Δεν είναι έτσι. Η διακυβέρνηση δεν είναι η διαρκής παρακολούθηση που θα καταστέλει. Είναι ένας χώρος εντό του οποίου πρέπει να φροντίσουμε ώστε το διαδίκτυο να προσφέρει ευκαιρίες σε όλους. Είμαι πεπισμένος για αυτό το στοιχείο και επίσης πεπισμένος είμαι ότι χρειάζεται να κάνουμε βήματα πρόοδου. Βεβαίως το Παγκόσμιο Φόρουμ ε, ε, ε, παρακολουθεί την νομοθεσία που προβλέπουμε. Σε ένα τόσο μεγάλο χώρο λοιπόν, τόσο ανεξέλεγκτο όπως το διαδίκτυο, δεν μπορεί να μην υπάρχουν σχετικές εξελίξεις. Ορθώς το έχουμε προβλέψει και ελπίζω να συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία, καθώς και το Ευρωκοινοβούλιο να διατηρήσει μια συνεπή στάση, μάλλον η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει μια συνεπή στάση, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ της Διακυβέρνησης για το διαδίκτυο. Και αυτό να ανανεώσει την εντολή του και να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπεθ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Να εκφραστώ και εγώ υπέρ της ανανέωσης της εντολής του Παγκόσμιου Φόρουμ για το διαδίκτυο και την ε, πολυσυμμετρική προσέγγιση. Απλώς να τονίσω εδώ μια σοβαρή πτυχή, την ανάγκη να βεβαιωθούμε ότι είναι ε, ελεύθερο και προσβατό σε όλους το διαδίκτυο. Πρέπει να φροντίσουμε την ουδετερότητα των δικτύων, να υπάρχει ελευθερία στην κυκλοφορία των πληροφοριών, ελευθερία στην έκφραση και να δώσουμε δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης. Ήδη έχουν καθοριστεί από την πλευρά του Πρόεδρου Ομπάμα σαφείς γραμμές για τη δημιουργία ακριβώς ε, ενός συστήματος προστασίας της ουδετερότητας. Τις τελευταίες ημέρες έχει προταθεί στους, ε, διακομετα... στους προμηθευτές να ε, λάβουν υπόψη αυτού του κανόνες για την τεχνολογική ουδετερότητα για ένα ανοιχτό και ελεύθερο διαδίκτυο, για την ελευθερία της έκφρασης και για να μπορέσει το δυναμικό καινοτομία να λειτουργήσει ελεύθερα και για την απασχόληση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Η διακυβέρνηση του δικτύου είναι ασφαλώ το ζήτημα του μέλλοντο. Η Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών έχει καταθέσει μία πρόταση η οποία αφορά τις, τις δραστηριότητες παρακολούθησης και στόχο έχει να αναλύσει τι είδους δυνατότητες προσφέρονται και διαπιστώνει ότι όχι μόνο μυστικέ υπηρεσίε μπορούν να αξιοποιήσουν αυτέ τι δυνατότητε παρακολούθηση. Είναι πάρα εύκολο ή πολύ σύντομα, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να εξασφαλιστεί η δυνατότητα για άλλες οργανώσεις ε, οποίες θα μπορούν να παρακολουθούν τη ε, διακίνηση στο διαδίκτυο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και τον ορισμό τη προστασία των συσκευών που χρησιμοποιούμε. Εγώ στη συσκευή την οποία χρησιμοποιώ θέλω να είμαι ο μόνος υπεύθυνο να αποφασίσω τι θέλω να ε, κυκλοφορεί, τι θέλω να ε, βγαίνει έξω από τον ε, ιδιωτικό μου χώρο, από την ιδιωτική μου σφαίρα. Πρέπει στο μέλλον δηλαδή να έχουμε τη δυνατότητα να ασφαλίζουμε επαρκώς τις συσκευέ που χρησιμοποιούμε, ώστε να μην μπορεί κανείς να μας καθοδηγεί. Να μην μπορεί κανεί εδώ την ώρα που βρίσκομαι εγώ μέσα στην Ολομέλεια να με καθοδηγεί και να μου κάνει σκόλο το χέρι μου από μακριά. Πρέπει να είναι ο πολίτη ασφαλής και βέβαιος ότι όπως εξασφαλίζεται το απόρριτο της αλληλογραφία, επί χάρτου θα εξασφαλίσετε και το απόρριτο της ε, ε διαγραμμικής του επικοινωνίας. Επίσης, Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε το δυναμικό που... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Σας διέκοψα. Δεν βλέπω την κυρία Φλεσικοβάβα Μπένοβα στην Ολομέλεια και έτσι καλώ την κυρία Σπυράκη. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Thank you, Mr. President. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Όχημα για να επιτευχθεί ο στόχος της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, της αγοράς που για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα ανοίξει σύμφωνα με εκτιμήσεις τις πόρτες σε πεντακόσια εκατομμύρια δυνάμει καταναλωτές, που μπορεί να αυξήσει το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ένωσης κατά 4% τα επόμενα δέκα χρόνια, περίπου 500 δισεκατομμύρια ευρώ. Και για το λόγο αυτό χρειάζεται το διαδίκτυο να έχει όσο το δυνατόν καλύτερη θεσμική υποστήριξη και κατοχύρωση μέσω μιας παγκόσμιας συμφωνίας κατοχύρωση για θέματα όπως είναι η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πολιτών όπως είναι η προστασία των παιδιών μας όπως είναι η ελευθερία του λόγου και η ελεύθερη διακίνηση των ιδεών. χρειάζεται υποστήριξη για ζητήματα ανοιχτά όπως η διαδικτυακή ουδετερότητα ώστε να διατηρηθεί το ανταγωνιστικό πεδίο για τις νέες καινοτόμες επιχειρήσεις που είναι αυτές που μπορούν να επαναφέρουν τη χαμένη ευρηματικότητα στην ψηφιακή τεχνολογία στο ευρωπαϊκό έδαφος. ως εκ τούτου το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου έχει από την πρώτη φορά που συνεδρίασε το 2006 στην ελλάδα συμβάλει πολύ θετικά στο διάλογο και την ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών αποτελεί ένα θεσμό που ενισχύει την αποτελεσματική κατάρτιση πολιτικής αναφορικά με το διαδίκτυο και γι' αυτό τάσσομαι υπέρ της ανανέωσης της εντολής του από το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο όχι μόνο γιατί θα πρέπει να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα στον οργανισμό ηνωμένων εθνών αλλά γιατί θα πρέπει μαζί και τώρα να ξεκινήσουμε να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα ώστε να ολοκληρώσουμε την τόσο σημαντική για την οικονομία μας ενιαία ψηφιακή αγορά αποχωρώντας, από τα εμπόδια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, κυρία Παούνοβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, Συζητάμε το ζήτημα της ανέωση εντολή του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Το διαδίκτυο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το εμπόριο τόσο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και εκτός. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο το διαδίκτυο επεκτείνεται εξαιτία ή χάρη μάλλον σε αυτό το πολύ θετικό μοντέλο διακυβέρνηση το οποίο υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά πανεπιστήμια, καθηγητέ, κυβερνήσει, μικρομεσαίε και μεγάλε επιχειρήσει που μπορούν και συμμετέχουν όλο και περισσότερο σε αυτό το νέο μοντέλο διακυβέρνηση του διαδικτύου. Θεωρούμε ότι έχει δημιουργηθεί το κατάλληλο πεδίο ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι το φόρουμ αυτό θα πρέπει να επεκταθεί, να συνεχιστεί περισσότερο. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει μία θετική προσέγγιση όσον αφορά τη διακυβέρνηση αυτήν και το 2015 μην ξεχνάμε ότι τα Ηνωμένα Έθνη θα αναθεωρήσουν τις γενικές πολιτικές που διέπουν αυτό το φόρουμ για τη διακυβέρνηση του δικτύου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε ένα μοντέλο, ένα πρότυπο ανοιχτού διαδικτύου, όπου θα έχουμε του απαραίτητου κανόνε όσον αφορά την περιαγωγή, όσον αφορά τα δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία. Πιστεύω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε πραγματικά να ολοκληρώσουμε την ενιαία ψηφιακή αγορά στην Ευρώπη. Σας ευχαριστούμε. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Υπάρχουν ορισμένοι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν ζητήσει ήδη το λόγο. Έχουμε τον απαραίτητο χρόνο στη θέσή μας αυτή τη φορά. Θα σας διαβάσω τα ονόματα των συναδέλφων που έχουν ζητήσει το λόγο με την ακόλουθη σειρά. Ε, Mr. Caputo, Mr. Marias, ε, Mr. Jakovcic, ε, Mr. Etheridge, Mr. Sojar, Madame Sojarova, Mr. Negrescu and Mr. Nagy and Mr. Boni. Και έτσι κλείνει ο κατάλογος. Κύριος Φανίστηλρόι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι που έχουμε πια αυτή την πρόταση τώρα από 7 χρόνια ψήφισμα και ευχαριστώ την πιλάρτα Καστίγιο και τους συναδέλφου τους άλλους. Αυτή λοιπόν η διάσκεψη, το φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών ε, αποτελεί τροφή για σκέψη αλλά και για το λιγότερο ανεπτυγμένο κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε και τη δική του συμμετοχή. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον Επίτροπο Άνσιπ. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει την μη κυβερνητική συμμετοχή εκπροσώπων του αναπτυσσόμενου κόσμου, γιατί ε, δεν θα προσφέρουν μόνο κυβερνήσεις κάποιες ιδέες, αλλά και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ας το σκεφτούμε αυτό. Εγώ έχω συμμετάσχει και στη διάσκεψη των Αθηνών και σε αυτή του Βίλνιους. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει όλη αυτή η επικοινωνία, η δυνατότητα επικοινωνίας με εκπροσώπους κρατών αλλά και μη κυβερνητικούς. Λυπούμε λοιπόν που έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Είναι κακό μήνυμα στην κοινότητα του διαδικτύου και γι' αυτό παρακαλώ να ξαναμπεί το θέμα αυτό στην ε, ημερήσια μας διάταξη. Ο Πρόεδρος ευχαριστώ πολύ και τώρα ο κύριος ε, Καπούτο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η ανανέωση της εντολής του Φόρουμ για την κυβέρνηση του δικτύου θα πρέπει να υποστηριχθεί από το Κοινοβούλιο μας. Από το 2005 το φόρουμ αυτό κατάφερε πραγματικά να προωθήσει ε, μια πολυμερή διαφανή συζήτηση όσον αφορά την κυβέρνηση του δικτύου και κατά αυτόν τον τρόπο αύξησε και τη δυνατότητα συνεργασία ε, τόσο τη κοινωνία των πολιτών όσο και των θεσμικών οργάνων. Το διαδίκτυο δραματίζει όλο και πιο σημαντικό ρόλο στη ζωή μα και παράλληλα με την άπτυξή του πρέπει να ασχοληθούμε με κάποια ζητήματα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, πώ θα προστατεύσουμε του ανήλικου που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, πώ θα καταφέρουμε να προωθήσουμε την ελευθερία τη έκφραση, τι θα κάνουμε το ζήτημα τη ιδιωτική ζωή, την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Νομίζω ότι Όλα αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη πόσο σφαιρικές είναι πλέον διασυνδέσεις στο διαδίκτυο, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει το φόρουμ αυτό και θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω του φόρουμ αυτού να καταφέρει να προωθήσει τις ευρωπαϊκές αρχές και τη συνεργασία μεταξύ θεσμικών οργάνων και κοινωνίας των πολιτών. Διακόπτει ο Πρόεδρος. Στόχος μας θα πρέπει να είναι να εγκινηθούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ένα ανοιχτό δίκτυο, ελεύθερο δίκτυο έκφρασης και διασύνδεσης μέσω διαδικτύου κύριε πρόεδρε το διαδίκτυο είναι γνωστό ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης και διευρύνει βεβαίως και τη δημοκρατία. τα ζητήματα όμως που πρέπει να αντιμετωπίσουμε είναι σημαντικά. τι κάνουμε με τα θέματα οικονομικής ισχύως διότι έχουν δημιουργηθεί μονοπωλιακές εταιρείες έχουν αποκτήσει δεσπόζουσα θέση πολλές φορές καταχρώνται αυτή τη δεσπόζουσα θέση ελέγχουν τις τεχνολογίες ελέγχουν την έρευνα παραβιάζουν τα ατομικά δικαιώματα το δεύτερο θέμα είναι επίσης ο ρόλος των κρατών. αυταρχικές κυβερνήσεις αποκλείουν την πρόσβαση στο διαδίκτυο περιορίζουν την ελευθερία έκφρασης παραβιάζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα παρακολουθούν τους ίδιους τους πολίτες. πρέπει λοιπόν να πάρουμε σοβαρά μέτρα να χτυπήσουμε την εγκληματική δράση που γίνεται μέσα από το διαδίκτυο να προστατεύσουμε την προσβολή της προσωπικότητας γι' αυτό λοιπόν το μοντέλο διακυβέρνηση πρέπει να είναι ανοιχτό πλουραλιστικό συμμετοχικό με την κοινωνία των πολιτών και τα πανεπιστήμια ασφαλές και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα. στηρίζω λοιπόν την ανανέωση της εντολής για το φόρουμ ε, που πρέπει να δώσει το κοινοβούλιο μα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το φόρουμ για την διακυβέρνηση του διαδικτύου είναι απαραίτητο. Επομένως ε, πρέπει να ανανεωθεί η θητεία του και όχι μόνο για ένα έτος. Εμείς θα θέλαμε να λάβει πιο μακροχρόνια εντολή, διότι θεωρούμε ότι έτσι θα είναι πιο αποτελεσματικό, θα λειτουργήσει καλύτερα. Θα ήθελα να τονίσω ωστόσο εδώ ότι όλες οι αρχές που αναφέρθηκαν, ελευθερία ανθρώπινα δικαιώματα, συνοδεύουν το διαδίκτυο μεν, όμως ε, δεν είναι μόνο μια υπηρεσία, ένα προϊόν σήμερα το διαδίκτυο, είναι ένας τρόπος ζωής. Ώρες είμαστε στο διαδίκτυο στη σημερινή εποχή. Δυστυχώ λιγότερο χρόνο περνάμε με τα αγαπημένα μας πρόσωπα και περισσότερο μπροστά στην οθόνη. Χρειάζεται μια νέα φιλοσοφία και γι' αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει την πέμπτη ελευθερία, την ψηφιακή ελευθερία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αρχίσουμε να τη συζητούμε γιατί αυτή η ελευθερία περιλαμβάνει και όλες τις αρχές αλλά και πολλούς κινδύνους. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Έθεριτς. Ευχαριστώ. Η μεγάλη δύναμη του διαδικτύου είναι ότι παρέχει ελεύθερα πληροφορίες σε όλους. Μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση ε, σε πάρα πολλές πληροφορίες ε, μέσα από ένα πολύ μικρό και φθηνό αντικείμενο συσκευή σε σχέση με το παρελθόν. Και σίγουρα πρέπει να ελέγχουμε και να ε, μπορούμε αυτή την ε, γνώση που είναι ελευθερία, που είναι δύναμη, να την προφυλάσσουμε από τις καταχρήσεις και σίγουρα όχι ε, να επιτρέψουμε την άνθηση του εγκλήματος μέσα από το διαδίκτυο. Ακόμη περισσότερο πρέπει να αποφύγουμε ότι οι πολιτικοί θα ελέγχουν το διαδίκτυο, την γνώση δηλαδή που προσφέρει. Οι πληροφορίες, οι γνώσεις πρέπει να ρέουν ελεύθερα μεν και ο άνθρωπος να μπορεί να έχει ε, επαφή και πρόσβαση στην αλήθεια και να γίνει μια δημοκρατική επανάσταση με την ελευθερία της έκφρασης και τη δημοκρατία που θα ισχύει για όλους. Και αυτή θα είναι μια μεγάλη μέρα όταν το πετύχουμε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σαϊρόβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, Σπάνια βλέπω να υπάρχει τέτοια σύμπνια σε όλο το πολιτικό φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτό γιατί αν συμφωνούμε, όπως ε, για το προκείμενο, θα μπορέσουμε να είμαστε και πρωταγωνιστές στο διεθνές προσκήνιο και για τη συζήτηση αυτού του θέματος, που είναι βέβαια η ανανέωση της ε, θητείας της εντολής του Φόρουμ για τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Όλοι θέλουμε να ανανεωθεί η θητεία αυτή. Και πραγματικά θα ήθελα όλοι οι βουλευτές να προωθήσουν ε, το ανοιχτό πνεύμα, την ε, ίση πρόσβαση και την αρχή της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, όπως βέβαια και της ε, ουδετερότητας του διαδικτύου. Επίσης, και άλλα σημαντικά, πολύ σημαντικά ζητήματα όπως είναι τα πνευματικά δικαιώματα, η ασφάλεια. Πρέπει να τα έχουμε υπόψη και ελπίζω οι εκπρόσωποι μας να υποστηρίξουν αυτές τις αρχές. Πρόεδρος κύριος Νικολέσκου. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Το διαδίκτυο θα πρέπει να είναι ελεύθερο. Θα πρέπει επίση να προστατεύονται οι χρήστε του διαδικτύου, καθώ επίση και όσοι αναπτύσσουν λογισμικό. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να βρεθεί στην πρώτη θέση της καταπολέμησης του εγκλήματος στο διαδίκτυο. Και γι' αυτόν τον λόγο θα πρέπει να συνεχίσουμε και την σημαντικότητα αυτή εντολή που έχει δοθεί στο Φόρουμ για την Κυβέρνηση του Διαδικτύου των Ηνωμένων Εθνών. Νομίζω ότι θα πρέπει να αντιταχθούμε σε διάφορες συμφωνίες όπως η συμφωνία της ΆΤΑ ή σε κάποιες προσπάθειες όπως αυτές που είδαμε στην Ουγγαρία προκειμένου να περιοριστεί η ελευθερία του διαδικτύου. Σαφώς χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο ασφάλειας και προστασίας, αλλά από την άλλη θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το διαδίκτυο αποτελεί ελπίδα δημοκρατίας για πάρα πολλούς ανθρώπους, ιδίως στις, ιδίως στις μη δημοκρατικές χώρες. Δίνεται επίση δυνατότητα στι μικρομεσαίες επιχειρήσει να επικοινωνούν μέσω διαδικτύου και επίση το διαδίκτυο δίνει την δυνατότητα σε απλού πολίτε να επικοινωνούν με τι οικογένειέ του, ιδίω όταν κατοικούν στο εξωτερικό. Ο κύριο Νάτσο έχει το λόγο. Η κατάσταση είναι τέτοια που το διαδίκτυο μπορεί να προσφέρει πολύ μεγάλη ανάπτυξη, μέχρι και 11%. Κατά 11% μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη. Ήδη στην οικονομία μας και αυτό το 11% μπορεί να αυξηθεί πολύ σύντομα κατά 5,7%. Ε, όφερος λοιπόν και για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για τους πολίτες. Η κοινότητα του διαδικτύου ενισχύεται όλο και περισσότερο. Είναι σημαντικό κομμάτι δηλαδή το διαδίκτυο της ζωής του καθενός μας. Αλλά βεβαίως η ελευθερία που προσφέρει δίνει πεδίο καταστρατήγησης και για πολλούς εγκληματίες ε, από εγκλήματα του κοινού ποινικού δικαίου, παραβίαση βασικών δικαιωμάτων σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών κτλ. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα καταπολεμήσουμε αποφασιστικά. Ευχαριστώ πολύ. Μπόνι. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Τέσσερα σημεία. Πρέπει να ανανεώσουμε την εντολή του φόρουμ για την ε, διακυβέρνηση του διαδικτύου Ευχαριστώ την Πιλάρ Καστίγια για την πρωτοβουλία. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό διότι βρισκόμαστε ενώπιον ε, μιας νέας μάχης για τις ε, θεμελιώδεις αξίες. Ελευθερία, ουδετερότητα του δικτύου, προστασία της θετικής σφαίρας. Δεν θέλουμε δηλαδή βαλκανοποίηση του διαδικτύου και μόνο μια Πολυμερή διαχείριση και διακυβέρνηση του διαδικτύου αποτελεί τη μόνη εγγύηση για την τήρηση των αξιών αυτών. Τρίτον, η πλατφόρμα που προσφέρεται για την συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο της εξισορρόπησης μεταξύ ελευθερίας, προστασίας του ιδιωτικού βίου, οικονομικής ανάπτυξης και ασφάλειας μέσω αυτού του φόρουμ είναι η καλύτερη δυνατή πλατφόρμα. Και τέταρτον, στην Ευρώπη χρειαζόμαστε πολύ πιο ε, σαφή διαρρύθμιση του δικτύου μεταξύ των διαφορών κέντρων συζητήσεως για το διαδικτύο. Ευχαριστώ. Κυρία Μορφάη, έχει το λόγο. Πρόεδρε, θα ήθελα να προτείνω να μιλήσουμε για τα ουσιαστικά θέματα. Απευθύνομαι προς τον Επίτροπο, λοιπόν. Και ρωτώ. Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με τη διερεύνηση παρακολούθηση. Διάφορες υπηρεσίες οι οποίες παρακολούν τους πολίτες παραβιάζοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν σε σχέση με όλες αυτές τις παραβιάσεις των ανθρώπινων δικαιωμάτων, παρακολουθήσει από τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά και άλλα κράτη που αναθέτουν στις υπηρεσίες τους ή και σε άλλους φορείς Πώς γίνεται, ποια είναι η κατασχέση με τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πριν από ένα χρόνο μόλις το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε έκθεση σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και καλό τον Επίτροπο να μας ενημερώσει για την πρόοδο των σχετικών ερευνών. Υπάρχει λοιπόν παρακολούθηση προσωπικών δεδομένων ακόμη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα, για να κλείσουμε τη συζήτηση, ο Επίτροπος Άνση. Κύριε Πρόεδρε, οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πολύ επικοδομητική αυτή συζήτηση. Ετέθησαν πολλά ζητήματα σήμερα και σε αυτά εστιάζουμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει το πολυσυμμετοχικό μοντέλο της διακυβέρνησης του διαδικτύου. Χάρη και στη συμμετοχή αυτής της κοινότητας, της πολυσυμμετοχικής κοινότητας στο διαδικτύο, με το διακρατικό πολυδιάστατο χαρακτήρα του κατάφερε να ανθίσει και να φέρει καινοτομία με όλα τα ωφέλη που αυτή συνεπάγεται για την ψηφιακή επανάσταση. Το φόρουμ συγκεντρώνει με επιτυχία διάφορους ευλεκόμενους ε, φορείς ε, και οι οποίοι συζητούν επικοδομητικά και αποτελεσματικά μεταξύ τους σε αυτά τα πλαίσια. Βέβαια πολλά μπορούν να γίνουν για να βελτιωθεί ακόμη περαιτέρω το δίκτυο καθότι είναι πολύτιμο, είναι ένα εργαλείο που βοηθά πολύ στη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Γνωρίζετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν από τους πιο σταθερούς ε, χρηματοδότες ε, και υποστηρικτές ε, του φόρουμ. Αυτό είναι ζωτικό για τη σταθερότητα που χρειάζεται αυτός ο οργανισμός για να λειτουργεί σωστά. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά όλος ιδιαίτερος και τη δική σας δουλειά Γενικά χρειάζεται πρόοδος ε, στη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Υπάρχουν δομές που πρέπει να περιλαμβάνουν τους πάντες, να είναι διαφανείς, ε, να έχουν την υποχρέωση της λογοδοσίας ε, και να τηρούν και τις σωστές τεχνικές προδιαγραφές. Η πόλη συμμετοχική διακυβέρνηση του διαδικτύου πρέπει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Πρέπει να είναι αξιόπιστο το διαδικτύο και να τους περιλαμβάνει όλους. Εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις αξίες της για το σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την πολυμορφία, τη διαφορετικότητα, το κράτος δικαίου, μπορεί να δείξει η ηγετική στάση εθνές επίπεδο. Θα πρέπει και μπορούμε να αρθούμε στο ύψος αυτού του καθήκοντος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντιπρόεδρε Άνσιπ. Έχω λάβει. Α, έχετε το λόγο για διαδικαστικό, κύριε Μορβάη. Ναι, δεν θα έπρεπε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι προφανές ότι ο κύριος Άνσιπ διάβασε κάτι που δεν ξέρω ποιος του έγραψε το πρώτο μισό αυτού του κειμένου το διάβασε στην αρχή και το δεύτερο μέρος μετά την υποτιθέμενη συζήτηση. Ως ε, πολιτικός που με έχουν εκλέξει μου θέλω να μου απαντήσετε στα ερωτήματα που σας έσαι κύριε Επιτροπή. Ο Πρόεδρος, δεν είναι ώρα των ερωτήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει την ελευθερία έκφρασης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αυτό το δικαίωμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν. Όπως έλεγα, έχω λάβει τέσσερις ε, προτάσεις ψηφίσματος με τις οποίες ολοκληρώνεται η συζήτηση.